Colleagues, may I ask you to take... Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. May I ask you the journalists to leave after... Θα ήθελα να ζητήσω από τους δημοσιογράφους να φύγουν ε, από εδώ μπροστά μετά από τα δύο πρώτα λεπτά όπου τους επιτρέπουμε να πάρουν κάποιες φωτογραφίες του υποψήφιου επίτροπου αλλά μετά τα δύο πρώτα λεπτά παρακαλώ θα πρέπει να Φύγετε από εδώ μπροστά μας, να φύγετε από αυτές τις θέσεις. Δύο ανακοινώσεις πριν να καλωσορίσω τον προσκεκλημένο μας. Θα ήθελα να ζητήσω από όσους παρακολουθούν την ακρόαση να μην κρατούν θέσεις που σαφώς φέρουν ονόματα άλλων και να σημειώσετε ότι η σημερινή διαδικασία μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει από το Γιάν 4Q1 την αίθουσα όπου μεταδίδεται η συζήτηση και επειδή υπήρξαν χειροκροτήματα στη διάρκεια κάποιων ακροάσεων, να θυμίσω ότι μόνο τα μέλη μπορούν να χειροκροτούν εάν το επιθυμούν. Uh, uh, και τώρα η κυρία Λουγκούσκοκ και εγώ θα συμπροεδρεύσουμε σύμφωνα με τη διαδικασία και να ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω τον υποψήφιο επίτροπο Βάλτης Δομπρόσκη σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική ακρόαση ενώπιον των δύο επιτροπών μας δηλαδή έκον και έμπλο. Όπως γνωρίζετε, ο στόχος της ακρόασης είναι να ασκήσει το δικαίωμά του το Κοινοβούλιο που απορρέει από τις συνθήκες να ψηφίσει για οποιοδήποτε ε, ομάδα επιτρέπων και ιδιαίτερα η ακρόαση των μεμονωμένων επιτρόπων απαιτούνται ώστε να αξιολογήσουμε τους υποψηφίους επιτρόπους επί τη βάση των γενικών τους ε, δυνατοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων, προσωπική τους ανεξαρτησία και ρεότητα, να, να, να αξιολογήσουμε τις επικοινωνιακές τους ικανότητες, τις πολιτικές τους προτεραιότητες, τις ικανότητες τους να αναλάβουν το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο και τη ε, συμφωνία τους με τις νέες προτεραιότητες της νέας Επιτροπής. Να θυμίσω πριν την ακρόαση ότι ο υποψήφιος ε, Επίτροπος είχε γράψει είχε απαντήσει γραπτό σε ένα προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο. Οι δε γραπτές του απαντήσεις έχουν διανεμηθεί σε όλες τις γλώσσες του ευρωβουλευτέ, και σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία ο υποψήφιος έχει υποβάλει και δήλωση συμφερόντων και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, είπε ότι δεν είχε καμία παρατήρηση όσον αφορά τη δήλωση συμφερόντων του υποψηφίου επιτρόπου. Η διάρθρωση αυτής της ε, συζήτησης ε, θα γίνει ως ήθιστε. Καταρχήν ε, θα έχουμε μια πρώτη εισαγωγική δήλωση του υποψηφίου επιτρόπου, όχι πάνω από 15 λεπτά. 5 λεπτά θα έχει επίσης ο υποψήφιος επίτροπος για μια τελική δήλωση και Εν τω μεταξύ θα έχουμε τρία, λεπτές ερωταπαντήσεις για τα μέλη. Ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση. Να θυμίσω επίσης ότι η αρχή των τριών λεπτών θα τηρηθεί αυστηρά, έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι οι συνάδελφοι να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους. Επίσης θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η διερμηνία παρέχεται από 23 γλώσσες, ώστε όλοι οι ομιλητές να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους και όπως είπα και σε άλλες ακροάσεις, θα σας ζητήσω να μην μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα, ώστε να μπορείτε, ε, ώστε να, μπορείτε να μεταφραστείτε από τους διερμηνείς. Επί της ουσίας τώρα, τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ο υποψήφιος επίτροπος Ντομπρόφσκης είναι πάρα πολύ κέρια, δηλαδή να καθοδηγήσει τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, να κάνει τη διακυβέρνησή μας πιο συνεπή, αποτελεσματική, δημοκρατική και να αντιμετωπίσει την σημερινή οικονομική κρίση, επιτυχάνοντας σταθερότητα την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ εργάζεται σκληρά για να παρέχει τη συμβολή του Κοινοβουλίου σε μια γνήσια ατζέντα για την ΟΝΕ και την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε την αναθεώρηση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης. Μαζί με εσά και τους άλλους υπεύθυνου επιτρόπους θέλουμε να εντοπίσουμε τον καλύτερο τρόπο και τη χρήση ε, του κανόνα της ευελιξίας ώστε να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στη σταθερότητα και στην ανάπτυξη για να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις και τις διαθετικές μεταρρυθμίσεις, να βελτιώσουμε την ε, οικονομική ε, τον συντονισμό και να αντιμετωπίσουμε τις υπάρχουσες διαφορές ανάμεσα στις αρμοδιότητες νομισματικής ε, πολιτικής και εκείνες ε, της οικονομικής πολιτικής και τέλος θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε και να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση μέσα στο πλαίσιο διακυβέρνησής μας. Αυτό το Κοινοβούλιο ζητά ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σύμφωνο. Και δίνω τώρα το λόγο στην Σύμπροέδρο Μαρίζα Ούσβολγκ για να συνεχίσει αυτή την εισήγηση. Ορισμένα σχόλια εξ Επιτροπής ε, απασχόληση και αυτό το κάνω στα σουηδικά, στη μητρική μου γλώσσα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο δυναμικό για να εγγυηθούμε την απασχόληση που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θα πρέπει να ορίσει αυτούς τους όρους για την προστασία των εργαζομένων. Χρειαζόμαστε μια κοινή αγορά που δεν θα πρέπει να μειώσει τις ε, καλές συνθήκες εργασίας ή να προβεί σε αθέμητο ανταγωνισμό, γιατί αυτό θα μπορούσε να επαπειλήσει και τις ε, συλλογικές συμβάσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διαχείριση της κρίσης στην αγορά εργασίας και θα πρέπει οι εταίροι να μπορούν να δράσουν αυτόνομα. Με την απόφαση Λαβάλ του δικαστηρίου βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο για την ελεύθερη κυκλοφορία. Επίσης υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν είναι σοβαρές και χρησιμοποιούν τα κενά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιούνκερ, στον ενακτήριο λόγο του μίλησε για την οδηγία περί αποσπασμένων εργαζομένων που θα πρέπει να επανεξεταστεί. Επίσης, αυτή η οδηγία θα πρέπει να αποτρέψει το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουμε τους ίδιους μισθούς για την ίδια εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν υπεύθυνοι για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο. Ο κύριος Ντομπρόφσκης θα είναι υπεύθυνος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει υποσχεθεί πολλά. Οι εταίροι θα πρέπει να προωθήσουν και το δικαίωμα διαπραγμάτευσης και θα πρέπει να προβλέπονται συγκεκριμένες δράσεις. Σε περίπτωση εκτροπών δεν μπορούμε να δεχτούμε μία άλλη οδό. Δεν μπορούν να ανταγωνίζονται τα κράτη-μέλη τα μεν τα δε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνουμε τώρα το λόγο στον